Buongiorno a tutti, possiamo cominciare. Chiedo scusa per questi pochi minuti di ritardo. Σας ευχαριστώ συνάδελφοι, πρέπει να ξεκινήσουμε αμέσως. Λοιπόν, ζητώ από όλους τους συνεργάτες να μας επιτρέψουν να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, η πρώτη ενημέρωση είναι τροποποίηση στην ημερήσια διάταξη Πολύ απλά θα σας ενημερώσω ότι το σημείο 20, αν δεν κάνω λάθος, το σχετικό με το feedback χειλή δεν θα συζητηθεί σήμερα για την αποστολή μας στη Χιλή λοιπόν τον Δεκέμβριο του 17 θα συζητηθεί τον μήνα Μάρτιο και όχι σήμερα ή αύριο. Τώρα για την ελεύθερη διαχείριση των μη προσωπικών δεδομένων θα δώσω αμέσως το λόγο στον εισηγητή μας. Έχει ε, τον λόγο ο συνάδελφος ο κύριος Κρανοντέψκι. Ευχαριστώ Πρόεδρε, είμαι ικανοποιημένος από την εξέλιξη των πραγμάτων. Η έκθεση αυτή από ό,τι φαίνεται δεν δημιουργεί αντιπαραθέσεις. Συνεπώς οι τροπολογίες ε, ακολουθούν νομίζω τον σωστή κατεύθυνση, ικανοποιούν τους συναδέλφους και με προσωπικά. Όλοι συμμεριζόμεθα τους ίδιους στόχους. Θα πρέπει να διασφαλίσουμε την ελεύθερη διακίνηση των δεδομένων στην Ευρώπη, των μη προσωπικών. Επαναλαμβάνω ότι πρόκειται για τα λεγόμενα mixed data, μεικτού τύπου δεδομένα. Και αυτό το λέω γιατί δημιουργούνται μερικές φορές ορισμένες ε, δυσκολίες κατανόησης. Θα πρέπει να ξεχωρίζουμε σωστά το ότι είναι προσωπικό δεδομένο, το τι είναι μη προσωπικό δεδομένο. Γενικά θα πρέπει να υπάρξει περαιτέρω ε, ευκρίνεια θα έλεγα στους χαρακτηρισμούς και να δούμε κάτω από και ποιες συνθήκες θα μπορέσουμε να εφαρμόσουμε τους συγκεκριμένους κανόνες. Ε, σχετικά με την ελεύθερη επαναλαμβάνω διακίνηση των δεδομένων. Έχουμε προτείνει ορισμένες λύσεις. Λέμε σαν παράδειγμα ότι όταν δεν μπορούμε να διαχωρίσουμε τα προσωπικά δεδομένα από τα μη προσωπικά, θα πρέπει να ε, έχουμε την δυνατότητα διάκρισης. Και το κείμενο πάνω στο οποίο εργαζόμαστε θα πρέπει να ε, ε, μας δίνει την δυνατότητα να χρησιμοποιούμε το GDPR με συστηματικό τρόπο. Ένα άλλο θέμα το οποίο συζητιέται με τους κοιόδης κυρίως στις είναι το τι μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έτσι ώστε να ελέγχονται σωστά οι ε, διαδικασίες και πράξεις εντοπισμού, γεωεντοπισμού. Εδώ θα πρέπει να τονίσω θετικά τις πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, ως προς το προκείμενο. Πρόκειται για συγκεντρωτική, επαναλαμβάνω, βάση δεδομένων και εδώ έχουμε προτείνει να υπάρξει ένα ενιοποιημένο πλαίσιο έτσι ώστε να μην υφίσταται η διασπορά των δεδομένων και τελικά για τη δημόσια διοίκηση θεωρούμε ότι και αυτή θα πρέπει να καλυφθεί από τις συγκεκριμένες προβλέψεις εφόσον διασυνδέεται με ατομικά υποκείμενα όταν προτείνονται ας πούμε υπηρεσίες προς τους πολίτες θα πρέπει να εντάσσεται στην ισχύ του κανονισμού. Ε, ε, φυσικά θα πρέπει να υπάρξουν εξαιρέσεις για θέματα δημοσίας ασφάλειας. Αυτά έχω πρόεδρε. Περιμένω ίσως πιθανές παρατηρήσεις και ερωτήσεις συναδέλφων. Ευχαριστώ. Ε, πάντως η έκθεση αυτή νομίζω δεν παρουσιάζει θέματα και πρέπει να υιοθετηθεί με ταχύτητα Έχω την αίσθηση ότι είναι αρκετά σημαντική έκθεση γιατί αποτελεί σημαντικό τμήμα της εσωτερικής αγοράς. Σας ευχαριστώ λοιπόν. Ε, δίνεται η δυνατότητα και στους σκιώδεις να πάρουν το λόγο η κυρία Ντικούνεν εξ του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστήσω και τον εισηγητή για το σχέδιο έκθεσης. Όπως γνωρίζουμε η δημιουργία της ενιαίας ψηφιακής αγοράς είναι βασικό σχέδιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα δεδομένα είναι μια σημαντική πτυχή. Οι ροές των δεδομένων είναι στην καρδιά των επιχειρησιακών ε, δραστηριοτήτων. Ε, όχι μόνο οι εταιρείε ε, πληροφορικής, αλλά και δημόσια διοίκηση, ηλεκτρικές υποδομές, γεωργία. Ε, η αξία της αγοράς δεδομένων εκτιμάται στα 60 δισεκατομμύρια ευρώ και θεωρούμε ότι θα φτάσει, θα ξεπεράσει τα 100 δισεκατομμύρια ευρώ το 2020. Είναι πολύ σημαντικό αυτό λοιπόν και για την ανάπτυξη και για την απασχόληση στην Ευρώπη αυτή η έκθεση σε ό,τι αφορά τα μη προσωπικά δεδομένα και την ελεύθερη ροή τους είναι εξαιρετικά σημαντική. Πρέπει να πάψουν να υπάρχουν ε, ε, υποχρεώσεις και απαιτήσει σε επίπεδο γεωντοπισμού, να απαγορευτούν αυτά για να βρεθούμε στο ίδιο επίπεδο με την Κίνα και τις ΗΠΑ. Συμφωνούμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι δεν πρέπει να υπάρχουν αχρίαστες εξαιρεσει. Θα πρέπει τα δεδομένα να ρέουν όσο γίνεται πιο ελεύθερα. Δεν πρέπει να υπάρχει επιπλέον επιβάρυνση για τις επιχειρήσεις που προσπαθούν να καινοτομήσουν στον τομέα της οικονομίας των δεδομένων. Όπως είπε ήδη ο εισηγητής, τα μεικτά αυτά δεδομένα είναι ένα θέμα το οποίο έχει αρχίσει να αναδεικνύεται. Εδώ πρέπει να βρεθεί μια λύση ε, που ε, να μην περιπλέκει περιπλέον τα πράγματα. Ήδη οι πολίτες και επιχειρήσεις δυσκολεύονται με την εφαρμογή του CDPR θα πρέπει λοιπόν να το εξετάσουμε το θέμα αυτό, διότι θα βρούμε μπροστά μας αυτά τα μεικτά δεδομένα και δεν είναι πάντα εύκολο να τα διαχωρίσουμε. Με τον εισηγητή και τους συνεισηγητές ε, θα επικεντρωθούμε στα ζητήματα αυτά τις επόμενες εβδομάδες με τους κοιόδης εισηγητές. Ε, θέλουμε λοιπόν ελεύθερη ροή δεδομένων στην Ευρώπη, είναι όμως ε, πολύ σημαντικό, ακόμα πιο σημαντικό, να δούμε πώς θα είναι πιο μεγάλη πρόσβαση στα δεδομένα αυτά. Είναι κάτι που συζητείται όλο και περισσότερο. Η πρόσβαση στα δεδομένα είναι εξαιρετικά σημαντική ε, για την καινοτομία, για τις επιχειρήσεις μας. Ε, χθες στην Επιτροπή Μεταφορών ε, εξετάσαμε την έκθεση πρωτοβουλίας του τομέα των μεταφορών και ζητήσαμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλει νομοθετικές προτάσεις σε ό,τι αφορά την πρόσβαση στα δεδομένα εντός των οχημάτων. Είναι αυτό πολύ σημαντικό για το σύνολο της ε, αλυσίδας αξίας, ε, αξιών ε, στην μηχανία. Είναι σημαντικό για το σύνολο του κλάδου στην Ευρώπη. Τα επόμενα βήματα λοιπόν είναι να ανοίξει, να ανοίξει η ροή δεδομένων στην ψηφιακή οικονομία. Θα ήταν καλό να μας πει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πώς σκοπεύει να προχωρήσει ε, σε ό,τι αφορά την ε, ανταλλαγή δεδομένων από επιχείρηση σε επιχείρηση. Είναι πολύ καλό ε, το σχέδιο κειμένου. Ευχαριστώ την εισηγητή. Είναι πολύ καλό σχέδιο για, ως βάση για περαιτέρω συζήτηση. Ευχαριστώ. Ο συνάδελφος Κόφατ δεν έχει έρθει ακόμα. Ο συνάδελφος ή συνάδελφος Κάλλας δεν μπορεί να είναι παρούσα. Ο επόμενος. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ τον εισηγητή, λέει ο κύριος Νταλούντε. Πράγματι θα πρέπει να δοθεί λύση στα θέματα χωρίς να δημιουργούνται προβλήματα με τα ε, γεωεντοπισμούς. Θα πρέπει να ανταλλάξουμε τις ε, βέλτιστες πρακτικές των κρατών μελών. Δεν θα πρέπει να καθορίσουμε όμως πάρα πολλές ε, εξαιρέσεις εμείς ανησυχούμε για την δυνατότητα χρήσης προσωπικών δεδομένων. Αυτά θα πρέπει να αποφασίζονται σε σχέση με το διαθέσιμο GDPR. Ένα άλλο θέμα το οποίο θα πρέπει να λαμβάνετε υπόψη είναι οι διοικητικές δυνατότητες των υπηρεσιών. Κάποια κράτη-μέλη θα α, ωφεληθούν από το ότι ο τομέας της πληροφορικής είναι πιο διαδεδομένος από ό,τι σε άλλους πέρα από τα θέματα γεωαντοπισμού, το vendor locking επίσης είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να αντιμετωπιστεί στο άμεσο μέλλον. Καλώς, Κάπελ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω για όλους του τις προσπάθειες ε, των εισηγητή, παρόλες τις ε, αρχικές διαφορετικές απόψεις. Σήμερα δεν υπάρχουν ε, πολλά αμφισβητούμενα ζητία. Πιστεύω πραγματικά ότι όσον αφορά τα δεδομένα στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να υιοθετήσουμε ένα μειογενές πλαίσιο. Τα στοιχεία αυτά και τα δεδομένα θα πρέπει με έναν συγκεκριμένο τρόπο και βεβαίως με κάποιους περιορισμούς απαραίτητους για την ροή των δεδομένων να μπορούν να μεταφερθούν. Σήμερα έχουμε συγκεκριμένες τεχνολογίες, γνωρίζουμε ποιοι είναι οι κίνδυνοι, γνωρίζουμε τις προπτικές τουλάχιστον λοιπόν μέχρι το 2020 μπορούμε να θέσουμε αυτό το πλαίσιο. Καταλαβαίνετε ότι έχει πολλαπλασιαστεί επί έξι η, ε, ο όγκος των δεδομένων. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό και εν ώψη των ποσών που διακυβεύονται, αλλά και του όγκου των δεδομένων, να έχουμε μια ελεύθερη ροή δεδομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι πολύ σημαντικό επίσης να λάβουμε υπόψη μας τις συγκεκριμένες παρατηρήσεις που έχουν γίνει για τους περιορισμούς. Και βεβαίως είναι σημαντικό οι εθνικές αρχές αλλά και οι ευρωπαϊκές αρχές να συντονιστούν και να υπάρχουν όταν υπάρχουν ε, ροές ε, που ξεφεύγουν από τα πλαίσια αυτά να μπορεί να υπάρχει εντοπισμός βάσει των σημερινών προδιαγραφών. Υπάρχει ο κώδικας συμπεριφοράς, ο οποίος θα πρέπει να εφαρμόζεται και οι εθνικές αρχές συνεχίζουν σήμερα να θέτουν περιορισμούς. Αυτοί οι περιορισμοί σε εθνικό επίπεδο θα πρέπει να πάψουν να εμποδίζουν τη ροή των δεδομένων. Γιατί μόνο με μια σωστή συνεργασία θα φτάσουμε στην πραγματική εφαρμογή αυτής, ε, αυτών των προτάσεων. Δεν υπάρχουν άλλοι σκιώδεις. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Και εγώ θέλω να πω ότι είναι ένα πολύ σημαντικό επόμενο βήμα όσον αφορά την ψηφιακή αγορά. Ξεκινήσαμε με το νομικό πλαίσιο που αφορά την περιαγωγή. Θέσαμε ήδη το πλαίσιο για την διασυνοριακή μεταφορά δεδομένων και με τη σημερινή μας πρόταση νομίζω ότι δυναμώνουμε ακόμα περισσότερο τις προσπάθειες συνεργασίας στον τομέα αυτό έχω την εντύπωση ότι όλοι οι αρμόδιοι οργανισμοί και φορείς ε, θα συνδράμουν. Υπάρχουν ακόμα θέματα που αφήνουμε για το μέλλον. Όλοι όμως ξέρουμε ότι η βάση για να υπάρχει μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα, καλύτερη επικοινωνία βάση των τεχνολογιών, οι οποίες βεβαίως διαρκώς ε, εξελίσσονται και σήμερα ξέρουμε ότι χρειάζονται τεχνολογίες και δυνατότητες οι οποίες να είναι όσον αφορά την ενεργειακή τους απόδοση πιο αποτελεσματικές, μία μεταφορά δεδομένων που να είναι πιο ασφαλής αλλά απρόσκοπτη. Και το ερώτημα τελικά είναι αυτό. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα πρέπει να μπορούμε να έχουμε τη δυνατότητα εντοπισμού και κοινοποίησεων όταν υπάρχουν ε, θέματα τα οποία δεν ε, εμπίπτουν στην πιστοποίηση ή όταν υπάρχουν πολύ νέες τεχνολογίες όπως ε, η οταν υπαρχουν πολλοι νεες τεχνολογιες οπως η τεχνολογια blockchain όπως ξέρετε, τους τελευταίους μήνες είχαμε εξαιρετικά θετικές εξελίξεις σε αυτό το νέο τεχνολογικό τομέα. Οι υπερυπολογιστές, super computing, θα πρέπει να στηριχθούν και σε κάθε περίπτωση στην Ευρώπη θα πρέπει να γίνουμε πρότυπο σε αυτό το τομέα. Θα δώσω το λόγο τώρα στον εκπρόσωπο της Γενικής Διεύθυνσης Connect της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Καλημέρα και να ευχαριστήσω τα αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τις εργασίες, τις τους για αυτό το σημαντικό φάκελο ό,τι αφορά την νέα ψηφιακή αγορά. Εμεί εκτιμούμε ιδιαίτερα το γεγονό ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει επιταχύνει τι εργασίε του για αυτό το σημαντικό ζήτημα μετά τη συμφωνία που επετέφθη στο επίπεδο Συμβουλίου το Δεκέμβριο επί του κειμένου που πρότεινε η Εσθονική Προεδρία. Σε ό,τι αφορά τώρα τα μεικτά δεδομένα, είναι ένα θέμα το οποίο θέτει και ο κλάδος. Πιστεύουμε ότι είναι σημαντικό οι κανόνε να είναι γίνεται πιο απλοί για τι επιχειρήσεις να είναι εύκολο δηλαδή να συμμορφωθούν με την ευρωπαϊκή νομοθεσία, ταυτόχρονα όμως να έχουμε τα κατάλληλα εχέγγυα σε ό,τι αφορά τα συγκεκριμένα δεδομένα. Η διάταξη για την ελεύθερη ροή στον κανονισμό αυτόν είναι απολύτως συνεπής με την, το νομοθέτημα GDPR. Έχουμε ένα νέο ε, πακέτο κανόνων που επιτρέπει την ελεύθερη ροή δεδομένων. Είναι λοιπόν ε, εντελώς νόμιμο να, για μια εταιρεία να επεξεργάζεται και να αποθηκεύει δεδομένα. Από εκεί και πέρα οι εταιρείε είναι αυτές που θα αξιολογήσουν πού είναι πιο ε, ε αποτελεσματικό και πού είναι πιο συμφέρον να γίνεται ο διαχωρισμός μεταξύ των προσωπικών και των προσωπικών δεδομένων το GDPR βεβαίως θα εφαρμόζεται για το προσωπικό σκέλος των δεδομένων, για τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και το, ε, τα λοιπά δεδομένα θα είναι ελεύθερης ροής. Βεβαίως οι υποχρεώσει τη προστασία δεδομένων ε, θα παραμείνουν για το σύνολο του πακέτου αν δεν μπορεί μπορεί να διαχωρίσει αυτά τα μεικτά δεδομένα. Είναι απολύτω ε, απαραίτητο να εξασφαλίσουμε πλήρη εφαρμογή του GDPR σε ό,τι αφορά τώρα την παρακολούθηση. Είναι πρόθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όντως να παρακολουθούμε ε, το πώς θα αναπτύσσονται οι διάφορες ε, ε, μέθοδοι ροής δεδομένων στην Ευρώπη. Ήδη η Ευρώπη είναι η Ήπειρος όπου λαμβάνουν χώρα μεγαλύτερες ροές. Όταν βλέπουμε ε, την ανταλλαγή μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση, τη ανταλλαγή μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και του υπόλοιπου κόσμου, είναι πολύ μεγαλύτερη ανταλλαγή, η ανταλλαγή δεδομένων εντό τη Ένωση από ότι με χώρε εκτό Ένωση ή από ότι η ε, ανταλλαγη ανταλλαγέ που λαμβάνουν χώρου μεταξύ άλλων περιφερειών εκτό Ευρώπη. Είμαστε λοιπόν ήδη στην πρώτη γραμμή σε ό,τι αφορά τη ροή δεδομένων και αυτό ο κανονισμό ε, θα βοηθήσει έτσι ώστε να επιταχύνουμε ε, αυτήν την τάση. Σε ό,τι αφορά τώρα την ενημέρωση όντως ε, πρέπει να υπάρχει, ε, να είναι απλή, να είναι εύκολη η πληροφόρηση της επιχειρήσης, ε, να έχουμε μία ενιαία δικτυακή πύλη. Γι' αυτό σκοπεύουμε λοιπόν να διαθέσουμε αυτές τις πληροφορίες έτσι ώστε να μπορούν οι επιχειρήσεις να τις χρησιμοποιήσουν εύκολα. Ενδεχομένως να υπάρχει και η νομοθεσία στην γλώσσα του εν λόγω κρατούς μέλους θα πρέπει αυτά τα στοιχεία να είναι διαθέσιμα και βάσει της εθνικής νομοθεσίας που θα μεταφέρει την Ευρωπαϊκή. Σε ό,τι αφορά τώρα την ανταλλαγή δεδομένων ε, μεταξύ επιχειρήσεων και αυτό είναι ένα σημαντικό στοιχείο τη οικονομία δεδομένων και τη ανάπτυξή Ήταν και βασικό στοιχείο τη ανακοίνωση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αν θυμάστε, τον Ιανουάριο πέρυσι για τη δημιουργία μιας ευρωπαϊκής οικονομίας δεδομένων, μπορώ να σας πω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, θα εγκρίνει ένα νέο ψηφιακό πακέτο την Άνοιξη και αυτό το πακέτο θα περιλαμβάνει μια σειρά από σημαντικά στοιχεία ε, για να προχωρήσει η οικονομία των δεδομένων. Μεταξύ άλλων και για την ανταλλαγή δεδομένων ε, μεταξύ επιχειρήσεων θα προκύψουν κατευθείαν γραμμές για αυτή την ανταλλαγή δεδομένων B2B ε, και θα, που θα καλύπτει και τα δεδομένα του δημόσιου τομέα. Επίσης ε, η Κομισιόν επεξεργάζεται την ανάπτυξη ενός κέντρου υποστήριξης για την ανταλλαγή δεδομένων ε, στα πλαίσια του B2B, δηλαδή της ανταλλαγής δεδομένων επιχείρηση με επιχείρηση. Ευχαριστώ την το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που εργάζεται από αυτού του σημαντικού φακέλου. Αναμένουμε επιτυχή έκβαση των προγραμματεύσεων όσο γίνεται πιο γρήγορα, έτσι ώστε να μπορέσει να ξεκινήσει ο τριμερής διάλογος ήδη επί Βουλγαρική Προεδρίας. Σας ευχαριστώ πολύ. Δεν ξέρω αν ο συνάδελφο Κρασνογιάσκη θέλει να απαντήσει, έχει το λόγο πάντω. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ήταν ε, εξαιρετικά χρήσιμα αυτά που ακούστηκαν. Ε, θα λάβουμε υπόψη μας τα στοιχεία αυτά. Να πω όμως ακόμα κάτι, αν μου το επιτρέπετε, για το πιο σημαντικό ζήτημα κατά την άποψή μου, τα μεικτά δεδομένα. Εμείς προτείνουμε μία λύση που θα μας επιτρέψει τα προσωπικά δεδομένα να περιλαμβάνονται όταν αυτά τα στοιχεία ε, ανταλλάσσονται για διοικητικούς σκοπούς και δεν είναι κάποια προσωπικά δεδομένα ε, απόρριτα. Ε, σε σχέση τώρα με την ε, λύση που ανέφερα ο συνάδελφος να αποφασίσουν τα δικαστήρια, ε, αυτό δεν θα ήταν καλό για τις μικρές επιχειρήσεις, για τις start-up. Το έχουμε ακούσει πολλάκι σε αυτό από τους εκπροσώπους του κλάδου. Βεβαίως θα τα εξετάσουμε όλα αυτά που ακούστηκαν σήμερα. Θα συνεχίσουμε λοιπόν να διαπραγματευόμαστε με τους συναδέλφους τους κοιόντες εισηγητές. Η τελευταία ενημέρωση για το θέμα αυτό μας λέει ότι η προθεσμία κατάθεσης των απολογιών είναι 27 Φεβρουαρίου. 16η απογευματινή, 18η απογευματινή, συγγνώμη. Περνάμε στο επόμενο θέμα πλαίσιο για τον έλεγχο των άμεσων εξωτερικών επενδύσεων, ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Δεν βλέπω όμως τον εισηγητή, ο οποίος από ό,τι μου είπαν έρχεται ο κύριος Μπούτι Κόφερ. Θα ήθελα να πω να ξεκινήσουμε με τους Κιώδης και όταν φτάσει ο εισηγητής θα πάρει το λόγο. Η κυρία Γκροστέτ για το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ο κύριος Μπουτικόφερ φτάνει. Madame Grosset è d'accordo, torniamo, riavvolgiamo il film e diamo la parola subito al rapporteur senza lasciargli... Να δώσουμε το λόγο στον εισηγητή, αφού έφτασε, ο κ. Μπουτικόφερ. Capito che si tratta di lui, sì. Monsieur Good morning, colleagues. Thank you. Καλή σας μέρα, αγαπητοί συνάδελφοι. Σας ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε την δυνατότητα να πω δύο λόγια για το θέμα αυτό στο οποίο καλούμεθα να συντάξουμε γνωμοδότηση Πρόκειται για ένα πλαίσιο που αφορά τις ε, επενδύσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχει ένα χρονοδιάγραμμα, το οποίο είναι γνωστό νομίζω στους συναδέλφους και δεν νομίζω ότι έχω να σχολιάσω κάτι από αυτού. Σε γενικές γραμμές, αν κοιτάξει κανείς αυτό το χρονοδιάγραμμα, αν θέλει κανείς να έχουμε αποτέλεσμα πριν το τέλος της θητείας, είναι εξαιρετικά ε, στενό, με την έννοια ότι το Κοινοβούλιο θα πρέπει να συμφωνήσουμε πριν το τέλος του χρόνου Αλλιώς δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει διαδικασία με το Συμβούλιο και να προλάβουμε να ε, προχωρήσουμε στην έγκριση. Το θέμα βεβαίως δεν είναι ένα θέμα επί του οποίου υπάρχει συνένευση, ξέρετε, της πρωτοβουλίας της Ιταλίας, Πολωνίας, Γαλλίας. Υπάρχουν όμως και χώρες που επιφυλάσσονται, που εκφράζουν ανησυχίες, όπως η Πορτογαλία. Η δική μου λοιπόν φιλοδοξία, δεδομένης της κατάστασης, είναι να υπάρξει ένας ε, μηχανισμός ε, επιλογής με την έννοια ότι θα ήθελα να υπάρξει επαρκής πλειοψηφία και εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά και βεβαίως ε, μεταξύ Συμβουλίου και Κοινοβουλίου στην τελική φάση της έγκρισης. Συμφωνώ με την επιλογή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μέθοδο εργασίας την οποία θεωρώ αποτελεσματική και περιγράφω την ε, πρόταση της Επιτροπής, ουσιαστικά δεν πρόκειται για μία ύπουλη, αν θέλετε, προσπάθεια να εισαγάγει προστατευτισμό από την πίσω πόρτα. Καθόλου. Καθόλου. Δεν υπάρχει τάση προστατευτισμού της ευρωπαϊκής βιομηχανίας εκτός από τις περιπτώσεις αυτές όπου υπάρχουν ε, υπόνοιες ότι αμφισβητείται η δημόσια τάξη και ασφάλεια. Πρόκειται λοιπόν για απλές προτάσεις και προσπαθούμε και εμείς με τις δικές μας προσθήκες να δημιουργήσουμε μια τέτοια πρόταση η οποία να είναι όσο λιγότερο γραφειοκρατική γίνεται, απλή. Σε κάποια σημεία λοιπόν που μου φαίνεται το κείμενο λίγο περίπλοκο, λίγο βαρύ, κάνω κάποιες προτάσεις εγώ έτσι ώστε να απλοποιηθεί λίγο το θέμα, να απλοποιήσουμε τις γραφειοκρατικές διαδικασίες και περιμένω τις ε, ε, αντιδράσεις σας για να δω αν αυτό βοηθάει ή αν υπονομεύει το πνεύμα του κειμένου. Πιστεύω ότι η σκοπός μας είναι να δημιουργήσουμε πραγματικές ευκαιρίες συνεργασίας, συνέργειας μεταξύ των κρατών μελών. Και βεβαίως σε καμία περίπτωση δεν θέλουμε να ασκήσουμε υπερβολική πίεση σε κάποιους από τους φορείς των κρατών μελών. Δεν θέλω δηλαδή κάποια κράτη-μέλη να υποχωρήσουν και να μην ε, συνεργαστούν ακριβώς επειδή θεωρούν ότι ε, υπάρχει υπερβολική πίεση από μέρους μας. Επαναλαμβάνω αυτό που έχω γράψει και στην ε, έκθεσή μου. Η απόφαση παραμένει και είναι καταρχήν μία απόφαση των κρατών μελών. Δεν υπάρχει ύπολη και κρυμμένη πρόθεση από μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να ε, σπρώξει κάτι. Αυτό είναι βασικό, αυτό είναι σαφές για μένα και μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορεί να υπάρξει συμφωνία. Οι προτάσεις μου νομίζω είναι σαφείς. Είμαι σίγουρος ότι όλοι τις διαβάσατε και μπορείτε να κάνετε τις παρατηρήσεις και τα σχόλιά σας. Κάτι θα ήθελα μόνο να πω που ίσως σας φανεί παράξενο όταν κοιτάξτε για πρώτη φορά το κείμενό μου. Είναι ο πιθανός ρόλος των συνδικαλιστικών οργανώσεων στην δημιουργία νομοθεσίας που αφορά τα εργασιακά θέματα. Πιστεύω ότι θα έπρεπε να δώσουμε έναν συγκεκριμένο και ε, καθοριστικό ρόλο στις συνδικαλιστικές οργανώσεις όταν θεωρούν ότι πλήττονται τα συμφέροντα των εργαζομένων. Κάποιοι θα με ρωτήσουν, μα γιατί δίνουμε τέτοια δύναμη, τέτοια εξουσία στις συνδικαλιστικές οργανώσεις. Θα σας εξηγήσω γιατί. Στις Ηνωμένε Πολιτείες υπάρχει μια τέτοια ιδέα που δίνει στα συνδικάτα τη δυνατότητα στις συνδικαλιστικές οργανώσεις να θίξουν, να αναφέρουν προβλήματα για οποιαδήποτε συμφωνία εμπορική είτε εάν θεωρούν ότι κάποιος εμπορικός εταίρος, κάποιος που συμμετέχει σε μια τέτοια ε, συμφωνία εμπορική, πλήττει τα συμφέροντά τους και εάν υπάρχει προσφυγή, όπως ξέρετε, από μέρους ε, κάποιου προς ε, έναν από τους εταίρους ε, αυτής της εμπορικής συμφωνίας, υπάρχουν στο τέλος, εάν καταδικαστεί ο συγκεκριμένος εμπορικός εταίρος, πολύ σημαντικές αποζημιώσεις. Γι' αυτό και επιτρέπει η αμερικανική νομοθεσία προσφυγή και από μέρους των συνδικαλιστικών οργανώσεων. Μπορούν λοιπόν οι εταιρείες να κρυφτούν πίσω από τις συνδικαλιστικές οργανώσεις και να ε, περάσουν κάποιες τέτοιες ε, προσφυγές, κάποιες τέτοιες διαμαρτυρίες από τη στιγμή που θεωρούν ότι θίγονται κάποια συμφέροντα. Νομίζω λοιπόν ότι είναι σαφές εδώ αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε, να είναι ξεκάθαρα τα πράγματα και σε καμία περίπτωση βέβαια να μην ε, υπονομεύουμε τα δικαιώματα και τη θέση των επιχειρήσεων. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ τον κύριο Μποτικόφερ. Έχει φτάσει ο συνάδελφος Σαβίνη και μετά η κυρία Γκροστέτ, αλλά πρώτα θα δώσω το λόγο στον κύριο Σαλίνη. Ευχαριστώ. Είχα τη δυνατότητα να συζητήσω και να ρίξω μια ματιά στα βασικά σημεία τα οποία θα χαρακτηρίζουν την θέση της ΣΥΤΡΕ για τον κανονισμό των συγκεκριμένων και όπως πολύ συχνά συμβαίνει στην αρχική φάση της ε, συζήτησης, ε, συμφωνούμε σε πάρα πολλά, ελπίζω να παραμείνει η συμφωνία αυτή. Θα πρέπει να πω ότι και η εισαγωγή την οποία έκανε ο κύριος Μπούτιχόφερ και η αρχική πρόταση την οποία έστειλε στους σκιώδους ε, δημιουργούν τις προϋποθέσεις σωστής εκκίνησης. Κάποιες παρατηρήσεις που ίσως να έχουν ήδη γίνει. Εγώ δεν άκουσα πλήρως την παρέμβαση του Κόφερα από ό,τι άκουσα όμως συμφωνούμε με την βασική γραμμή η οποία λέγει ότι είναι σωστό, αν και ακούγεται λίγο ρητορικό, να υπογραμμίσει κανείς ότι για τον έλεγχο των εξωτερικών άμεσων επενδύσεων εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν σημαίνει νέες μορφές προστατευτισμού Σημαίνει όμως ότι θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε κάτι το καινούριο, ότι δηλαδή οι επενδύσεις σε ένα συγκεκριμένο κράτος μέλος επηρεάζουν και τις υπόλοιπες χώρες. Το θέμα είναι λοιπόν πώς θα μπορέσουμε να εκινήσουμε μία μορφή εναρμονισμού της στρατηγικής επενδύσεων που να επηρεάζει θετικά όλες τις χώρες σαν παράδειγμα μια επένδυση στον Πειραιά επηρεάζει την Γαλλία, την Ιταλία κτλ. Συνεπώς λοιπόν το βασικό μας θέμα είναι και μιας και σήμερα μόνο 12 από τις 27 χώρες έχουν συστήματα ελέγχου επί των άμεσων επενδύσεων να προσπαθήσουμε να δώσουμε κίνητρα για να υπάρξει μια ενιαία αντιμετώπιση από όλες τις χώρες έτσι ώστε ο έλεγχος αυτός να γίνεται από όλες τις χώρες μέλη και είναι σωστή η ε, διαπίστωση σύμφωνα με την οποία η αρμοδιότητα ε, παραμένει αρμοδιότητα εθνική. Εμείς δεν θέλουμε να ανακατανύμουμε μια παραδοσιακή αρμοδιότητα εθνικού τύπου. Θέλουμε διατηρώντας την αρμοδιότητα αυτή να δούμε ακριβώς ποιες είναι οι επενδύσεις των άμεσων ξένων επενδύσεων και πώς επηρεάζουν το σύνολο της Ένωσης. Ένα δεύτερο σημαντικό στοιχείο είναι ότι για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε ένα αποτελεσματικό σύστημα ελέγχου θα πρέπει να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις έτσι ώστε τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται στον έλεγχο αυτό να συμμερίζονται και οι πιθανές χώρες επενδυτές εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν θέλουμε εμείς να έχουμε συστήματα ελέγχου εάν δεν είναι καρπός ενός μηχανισμού αμοιβαιότητας. Δεν θα μπω τώρα στην ουσία των μεμονωμένων τροπολογιών όπως έκανε ε, ο εισηγητής γιατί δεν είναι αυτή η σωστή συγκυρία. Αλλά νομίζω ότι γενικά ε, πρέπει να συμφωνήσουμε με πολλά από αυτά και μία παρατήρηση για την ανάλυση που έκανε ο Μπούτικο τη συμμετοχή των συνδικαλιστικών οργανώσεων είναι θέμα σημαντικό προς και πράγματι όταν βλέπουμε τι συμβαίνει στι Ηνωμένε Πολιτείε, το θέμα αυτό είναι σημαντικό, δεν θα πρέπει να παραμείνει θεωρητικό. Γνωρίζουμε ότι οι σχέσεις ανάμεσα στην χώρο της οικονομίας και τις συνδικαλιστικές οργανώσεις στην Ευρώπη είναι καρπός θα έλεγα κάποιων συνδικαλιστικών χαρακτηριστικών στην Ευρώπη ε, εντελώς διαφορετικών από τα αμερικανικά unions Προϋπόθεση λοιπόν για να εφαρμοστεί αυτό το οποίο ζητά ο εισηγητής σημαίνει ότι θα πρέπει να υπάρξει μια πολύ σημαντική τροποποίηση του τρόπου λειτουργίας των συνδικαλιστικών οργανώσεων και της ε, διάρθρωσης των νομικών ρυθμίσεων για τα εργασιακά, ιδιαίτερα στη χώρα μου. Πάντως γενικά πάμε καλά. Θα δώσω τώρα με χαρά τον λόγο στον συνάδελφο Μαχτά, σοσιαλιστές. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Να πω καταρχήν κάποια γενικότερα, κάποια γενικότερα σχάλια, σχόλια. Ο 20ος αιώνας ήταν διπολικός, αλλά ο 21ος θα είναι σίγουρα πολυπολικός και σε επίπεδο ασφάλειας ε, ε δεν είναι οι ίδιοι πλέον οι εταίροι μα. Ε, αυτό δεν ισχύει μόνο για την Ευρωπαϊκή Ένωση, ισχύει και για το κάθε κράτο μέλο. Έτσι όπω το βλέπω εγώ λοιπόν, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να εγκαταλείψει αυτήν την α, αγαθή έτσι, αποδοχή των ξένων επενδύσεων. Είμαστε οι μόνοι που δεν έχουμε ένα σύστημα φιλτραρίσματος. Ενώ στην Κίνα, στην Αυστραλία, στι ΗΠΑ έχουν ενισχύσει του ελέγχου των ξένων επενδύσεων. Δεν μπορούμε λοιπόν εμείς να είμαστε η αγαθή του παγκόσμιου χωριού. Οι επενδύσεις από ε, υπηκόους τρίτων χωρών ανταγωνιστικών προς την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι κάτι που πρέπει να μας προβληματίσει. Δεν πρέπει να εξαρτώμεθα ούτε τεχνολογικά ούτε οικονομικά. Πρέπει να έχουμε μια στρατηγική ανεξαρτησία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της. Διότι ιδάλλως θα είμαστε ευάλωτοι τα συστήματά μας, τα δίκτυά μας θα είναι βάλωτα. Μιλάμε για πολύ σημαντικούς ε, παράγοντες ε, ε, διάδοσης απειλών, όπως η ΙΗ. Συμφωνώ με πολλέ προτάσει του εισηγητή, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τον ενεργό ρόλο των, των συνδικάτων, ο ενισχυμένο ρόλο του, του, του Κοινοβουλίου, ο ευρωπαϊκό χαρακτήρα των συστημάτων και η ενίσχυση του συντονισμού ε, των μηχανισμών φιλτραρίσματος. Όμως ε, θέλω να πάω ακόμα παραπέρα. Ε, θα ήταν εύκολο να κρατήσουμε μια αμυντική στάση και να ε, υπερασπιστούμε το status quo. Θα μπορούσαμε να πούμε εμείς στη Γαλλία ότι δεν πρέπει ο μηχανισμός φιλτραρίσματος ο δικός μας ε, να επηρεαστεί από αυτό τον κανονισμό. Όμως έχουμε τώρα περισσότερα δίκτυα, έχουμε ροές, έχουμε ε, διάδοση των κινδύνων. Ε, η κάθε αλυσίδα είναι όσο ισχυρή, ισχυρό είναι ο πιο δύναμος κρίκος της και αυτό είναι, πιο, είναι αληθινό περισσότερο από ποτέ σήμερα. Πέρα λοιπόν από το δυνητικό χαρακτήρα του φιλτραρίσματος όπως προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, δεν μπορεί να έχουμε απλά ένα κατάλογο βέλτιστων πρακτικών. Πρέπει να ενισχύσουμε το μηχανισμό που θα μπορεί να ενεργοποιήσει η Κομισιόν βασιζόμενη στην ομάδα που προτείνει ο εισηγητής ε, ταυτόχρονα όμως αυτό θα πρέπει να το διαβρύνουμε σε όλα τα κράτη-μέλη και στα κράτη-μέλη εκείνα που δεν έχουν κανένα σύστημα φιλτραρίσματο. Τέλος, για τα, για τα κριτήρια και τους διάφορους τομεί δεν έχει επιληθεί ακόμα, δεν έχει κλείσει η συζήτηση αυτή. Πρέπει να αποφασίσουμε. Θα πρέπει επίσης η προθεσμία για τι ε, ε, ε, να πάει μία εβδομάδα πίσω, διότι η Επιτροπή Ίντα έχει ένα χρονοδιάγραμμα πιο μεγάλο, πιο μακρύ, 26 Μαρτίου αν δεν κάνω λάθος. Θα έλεγα λοιπόν και εμείς να πάμε μια εβδομάδα πιο πίσω την προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών. Νομίζω ότι είναι εύλογο το αίτημά σα. Θα μας πει ο εισηγητής την άποψή του για το χρονοδιάγραμμα. Αυτό πράγματι θα επιτρέψει να εμβαθύνουμε καλύτερα στο θέμα ε, δεν βλέπω τον σκιώδη των συντηρητικών. Φτάνουμε στην κούε λοιπόν. Λόπες Βεμέχο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω και τον εισηγητή για την παρέμβασή του. Λοιπόν, ε, έχουμε διάφορα ερωτήματα εδώ. Πρώτον, είναι προφανές ότι είναι αναγκαίο να υπάρχει έλεγχος των άμεσων επενδύσεων στις τρίτες χώρες. Αυτό αιτιολογείται, το καταλαβαίνουμε, τα κράτη-μέλη και η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να το αναλάβουν αυτό. Ε, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα από αυτού. Εκεί όμως που υπάρχει πρόβλημα με αυτές τις επενδύσεις χωρί όρια ε, όπου ο καθένα μπορεί να κάνει ό,τι θέλει μπορεί να χαθούν ε, θέσεις απασχόλησης. Μπορεί δηλαδή να επιδεινωθεί το επίπεδο ζωής των Ευρωπαίων. Εάν δεν ελέγχουμε αυτές τις επενδύσεις υπάρχουν και κίνδυνοι αν, ζημίας ανεπανόρθωτης ε, για το περιβάλλον. Διαπιστώνουμε ότι τα κράτη-μέλη και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορούν να ελέγχουν τι είδους ξένες επενδύσεις μπορούν να γίνουν αποδεκτές και ποιε όχι σε άλλα κράτη-μέλη. Αυτό θέλουμε εμείς. Θα πρέπει να υπάρχει ένα δικαίωμα βέτο από τη μία χώρα προς την άλλη σε ό,τι αφορά τις συγκεκριμένε επενδύσεις. Εμείς συμφωνούμε με την ανταλλαγή πληροφοριών. Εκεί όμως που δεν συμφωνούμε είναι να υπάρχει μια απέτηση εξήγηση, ή ένα άμεσο βέτο ε, για, για ένα άμεσο βέτο σε μια επένδυση. Ιδιαίτερα όταν αυτό βασίζεται σε ε, επιχειρήματα δημόσιας τάξης και ασφάλειας ε, που μπορεί να χρησιμοποιηθούν αρκετά αυθαίρετα ε, κάποιοι είναι εχθροί, κάποιοι είναι φίλοι, δέχονται αυτές τις επενδύσεις, κάποιοι άλλοι δεν τις δέχονται, ενώ στην πραγματικότητα είναι οικονομικοί οι λόγοι και δεν έχω καμία σχέση με την ασφάλεια ή τη δημόσια τάξη. Εμείς θεωρούμε ότι θα πρέπει να αναλυθούν κάποια από τα στοιχεία που έχω προταθεί εδώ, χρειαζόμαστε χρόνο. Συμφωνούμε λοιπόν να παραταθεί η προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών για να μπορέσουμε να εξετάσουμε ενδελεχέστερα τα διάφορα στοιχεία και επίσης συμφωνούμε και συμφωνούμε και με τον εισηγητή εδώ ότι ο ρόλος των συνδικαλιστικών οργανώσεων θα πρέπει να είναι πιο ενεργός θα πρέπει πραγματικά να παίζουν ένα σημαντικό ε, ρόλο κατά τη λήψη αποφάσεων θα συνεχίσουμε εμείς τις εργασίες μας. Ε, από εκεί και πέρα αυτό που έχει σημασία για μας, όπως είπα, δεν είναι ότι οι πληροφορίες οι ίδιες ε, που πρέπει να κυκλοφορούν προφανώς, αλλά πρέπει μια χώρα να μπορεί να αποφασίσει ε, ε να, να μην, να μπορεί να αποφασίσει για τις επενδύσεις μιας άλλης χώρας. Δεν υπάρχει λοιπόν των φιλελευθέρων και του NRF ε, ε, ο Σκιώδης, οπότε περνώ στους μεμονωμένους ε, ομιλητές. Ρούμπιχ. Ευχαριστώ πολύ. Όντως είναι πολύ σημαντικό το θέμα, γιατί οι επενδύσεις δημιουργούν θέσεις απασχόλησης. Είναι πάντα καλές οι επενδύσεις για τις για την ανάπτυξη, τουλάχιστον εάν χρησιμοποιούνται και κατευθύνονται προς την σωστή κατεύθυνση. Βεβαίως υπάρχουν και θέματα προστασίας των επενδύσεων, είναι το θέμα της αμοιβαιότητας, αυτό ψάχνουμε, ισορροπημένη δηλαδή προσέγγιση και να υπάρχει ίση μεταχείριση των επιχειρήσεων αυτών που ήδη υπάρχουν και επενδύουν και δραστηριοποιούνται στη συγκεκριμένη χώρα. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει η νομική δυνατότητα προστασίας όλων αυτών των ήδη υπαρχουσών επενδύσεων και επιχειρήσεων. Με προσοχή Θεωρώ ότι η συνεργασία με τα τρίτα κράτη σαφώς και θα πρέπει να περάσει μέσα από αυτήν την πρόταση. Έχουμε και τον συγκεκριμένο χάρτη για τις επενδύσεις ε, σε μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτων χωρών. Αυτό θα πρέπει σαφώς να υπογραφεί από περισσότερες χώρες η ανάπτυξη περνάει μέσα από αυτές τις επενδύσεις και είναι απαραίτητη η διευθέτηση αυτού του νομικού πλαισίου. Η κυρία Γκροστέτ. Ευχαριστώ. Κυρία Πρόεδρε, ευχαριστούμε νομίζω τον εισηγητή για την εργασία του. Όντως, το θέμα των ε, επενδύσεων, των ξένων επενδύσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η επιλογή τους, ε, το screening που πρέπει να γίνεται σίγουρα είναι κάτι το πάρα πολύ σημαντικό. Ένας ευρωπαϊκός έλεγχος δηλαδή. Εννοείται ότι είναι πολύ σημαντικό να μπορούμε να προσελκύσουμε επενδύσεις ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι μια ευκαιρία για την οικονομία μας, αλλά θα πρέπει να μπορούμε να επιλέγουμε και να ελέγχουμε αυτές τις επενδύσεις. Από τη στιγμή δηλαδή που γίνεται η επιλογή, που επιβεβαιώνεται η δυνατότητα για μια επιχείρηση να επενδύσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα πρέπει να συνεχίσουμε την παρακολούθηση καθότι μία ξένη επένδυση σε καμία περίπτωση δεν θα μπορεί ανεξέλεγκτα από εκεί και πέρα να κάνει ε, οτιδήποτε επιλέγει. Δεν δίνουμε δηλαδή μία εν λευκό επιταγή στις ξένες επιχειρήσεις να επενδύσουν στην Ευρωπαϊκή Έπτωση. Θα πρέπει να συνεχίσουμε να παρακολουθούμε. Ευχαριστώ πολύ και δίνω το λόγο στην εκπρόσωπο της DigiTrade. Παρακαλώ ε, να είσαστε αρκετά συνοπτικοί και πλησιάζει η ώρα των ψηφοφοριών. Δεν έχουμε χρόνο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ τα μέλη της Επιτροπής, ευχαριστώ τον εισηγητή για την υποστήριξή του και για τις παρεμβάσεις που ακούστηκαν προηγουμένως και δείχνουν ότι υπάρχει πραγματικά στήριξη για την συγκεκριμένη πρόταση που κατέθεσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την οποία θεωρούμε πράγματι ανάλογη με τις προσπάθειες και τα μέσα που έχουμε. Να αναφερθώ σε, σε κάποια σημεία τα οποία παρατηρώ στις προτινόμενες τροπολογίες γιατί αν θα υπάρχει δυνατότητα σχολιασμού σε προγραμματισμένες και ολοκληρωμένες μορφές επενδύσεων το είπε και η τελευταία ομιλήτρια. Η τροπολογία προτείνει οι γνωμοδοτήσεις αυτές να γίνονται για προγραμματισμένες επενδύσεις. Νομίζω να, ότι πρέπει να τονίσουμε ότι υπάρχουν μηχανισμοί screening στην Ευρώπη που δίνουν την δυνατότητα να εκφραστούν απόψεις και για ολοκληρωμένες μορφές επένδυσης. Πιστεύουμε επίσης ότι έχει νόημα να υπάρχει δυνατότητα αντιμετώπισης πιθανών θεμάτων στον τομέα της ασφάλειας, ε, τα οποία αντιλαμβανόμεθα και διαπιστώνουμε εκ των υστέρων. Να υπάρχει δηλαδή δυνατότητα για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα κρατημέλη να υπογραμμίζουν τους κινδύνους και να προτείνουν αντίμετρα, ε, ακόμα και αν οι επενδύσεις αυτές έχουν πλέον ολοκληρωθεί και να μην παραμείνουμε μόνο στην προγραμματική φάση. Το δεύτερο σημείο είναι η υποχρέωση δημοσιοποίησης Κατανοούμε τις προθέσεις του κυρίου Μπουτικόφερ να μειωθεί το γραφειοκρατικό άχθος και είναι κάτι το οποίο μας βρίσκει σύμφωνος. Εμείς έχουμε προτείνει ένα σύστημα το οποίο απαιτεί ε, το ελάχιστο επίπεδο ανταλλαγής πληροφοριών αλλά ουσιαστικό επίπεδο πληροφοριών έτσι ώστε να μπορέσει να λειτουργήσει το σύστημα τέλος η συζήτηση για την συστηματική μορφή ελέγχου των προγραμμάτων ευρωπαϊκού χαρακτήρα και συμφέροντος. Εμείς δεν στοχεύουμε ένα σύστημα το οποίο να απαιτεί συστηματικό έλεγχο κάθε επένδυσης ξεχωριστά. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα απαιτήσει μια γραφειοκρατική ομάδα την οποία δεν θα θέλαμε να δημιουργήσουμε εμείς, θα θέλαμε να περιορίσουμε τους έλεγχους μόνον σε συγκεκριμένες περιπτώσεις στις οποίες παρουσιάζονται κίνδυνοι για την ασφάλεια και όχι σε συστηματική μάλιστα βάση. Και γι' αυτό ακριβώς θα θέλαμε και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας δώσει την δυνατότητα να κάνουμε ένα screening και όχι να επιβάλλουμε ένα συστηματικό μηχανισμό. Και τέλος για το θέμα των συνδικάτων είναι σαφές ότι πράγματι στο Ηνωμένο Βασίλειο το εμπόριο στα πλαίσια των εμπορικών συμφωνιών τα συνδικάτα παίζουν ένα σημαντικό ρόλο ε, να θυμίσω ότι ο έλεγχος, ε, ε, στον έλεγχο, το screening, το screening που γίνεται στις Ηνωμένες Πολιτείες για ξένες επενδύσεις, η δυνατότητα αυτή δεν προβλέπεται για τα συνδικάτα. Μιλάμε όχι γενικά για τα συμφέροντα των συνδικάτων, αλλά για θέματα ασφαλείας. Ο κύριος Μπούτικοφερ, αν θέλει να κλείσει τη συζήτηση στην παρούσα φάση. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ και όλους τους συναδέλφους που πήραν το λόγο. Για μένα είναι εντελώς αποδεκτά αυτά που ζητάτε, τουλάχιστον ε, όπως πρότεινε ο κύριος Μαχτά να επιμηκυνθεί κατά μία εβδομάδα. Δεν έχω απολύτως καλέλα πρόβλημα για την υποβολή των τροπολογιών η προθεσμία. Επίσης άκουσα αυτό που είπατε, την ανησυχία σας δηλαδή, ότι κάποιες χώρες θα μπορούσαν, επειδή έχουν κάποιες επιφυλάξεις ή αντιρρήσεις, να εμποδίσουν με βέτο την όλη διαδικασία. Αυτό που φοβάμαι όμως και αυτό που θέλω να αποφύγω είναι καταχρήσεις αυτού του δικαιώματος. Και θα πρέπει πραγματικά να προσπαθήσουμε να αποφύγουμε ιεραρχικές σχέσεις μεταξύ των κρατών μελών. Και αυτό που προτείνει η Επιτροπή, δηλαδή έναν εκ των ε, έλεγχο, έναν μια εκ των υστέρων δυνατότητα ε, αντίρρησης, αυτό έχουμε χρόνο να το συζητήσουμε. Από τη στιγμή που μιλάμε όμως για ένα μηχανισμό screening, επιλογής, ελέγχου δηλαδή, από τη στιγμή που έχουμε ένα κανονισμό ο οποίος ουσιαστικά προβλέπει όλες αυτές τις δυνατότητες ελέγχου και επιλογής, δεν μπορούμε να πούμε ότι και εξ δηλαδή εκ των υστέρων γίνεται ανταλλαγή πληροφοριών που ουσιαστικά δεν θα επηρεάσει όμως καθόλου την απόφαση. Απλώς αποδεικνύω πόσο αδύναμος είμαι, πόσο δύσκολο είναι για μένα να επηρεάσω τα πράγματα. Για μένα αυτό πραγματικά δεν πρέπει να το κάνουμε. Και το θεωρώ και αντιπαραγωγικό αλλά και λάθος, ε, θεωρητικά λάθος. Τώρα, όσον αφορά τις λεγόμενες στρατηγικές επενδύσεις, τις στρατηγικές υποδομές και δεν αναφέρομαι μόνο στο νερό, στα δίκτυα της ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά και παραδείγματο χάρη η πολυμορφία των μέσων. Και αυτό αποτελεί για μένα μια στρατηγική υποδομή. Στην Τσεχία, παραδείγματο χάρη, βλέπουμε κάποιους ε, προσπάθειες ε, να υπάρξει επέμβαση από μέρους κάποιων Κινέζων ή άλλων παραδείγματος χάρη στην εσωτερική πολιτική της Τσεχίας. Αυτό βάσει του Αμερικανικού νόμου δεν θα μπορούσε να είχε γίνει. Θα ήθελα λοιπόν πραγματικά όλες οι επενδύσεις βεβαίως ε, κατά κάποιο τρόπο να παρακολουθούνται, αλλά κυρίως, κυρίως να ελέγχονται οι επενδύσεις αυτές που θα μπορούσαν να απειλήσουν αυτές τις καθοριστικές ε, ελευθερίες, ε, την ασφάλεια, τη δημόσια τάξη, καθοριστικές για την Ευρώπη. Και γι' αυτό και πραγματικά επιμένω σε αυτό το θέμα νομίζω των συνδικαλιστικών οργανώσεων, το εξήγησα αρκετά. Η συζήτηση ήταν ενδιαφέρουσα, τελειώσαμε λοιπόν με το κομμάτι ε, για τη συζήτηση πριν της ψηφοφορίες, συμπερασματικά πάντως και σχετικά με την κατάθεση των τροπολογιών. Ο εισηγητής είναι διαθέσιμος με το έτοιμά σας. Νομίζω ότι και οι υπόλοιποι συνάδελφοι θα συμφωνήσουν. Να αφήσουμε λοιπόν στην Γραμματεία και το Προεδρείο ε, να συμφωνήσουν για την κατάθεση των τροπολογιών. Θα σας ενημερώσουμε το ταχύτερο δυνατόν. Έρχεται ο πρόεδρος Μπούζεκ για να ξεκινήσουμε και τις ψηφοφορίες. Richard had the same idea. Uh, good morning, dear colleagues. Dear morning. Αγαπητοί συνάδελφοι, καλή σας μέρα. Αγαπητοί συνάδελφοι, αποφασίζω τον Αντιπρόεδρο, τον κύριο Χάνκελ, ε, την Αντιπρόεδρο μάλλον. Δεν ήταν ο κύριος Χάνκελ. Α, ήταν η κυρία Τόιερ. Α, συγγνώμη. Πού είναι η κυρία Τόιερ. Ε, κάποιος μου είπε ότι ήταν ο κύριος Χένκελ. Η πρώτη αντιπρόεδρος, η κυρία Τόιερ, είναι εδώ μαζί μας. Ε, όχι ακόμα. Εν πάση περιπτώσει, εγώ είμαι ευγνώμων στην κυρία Τόιερ που ε, προείδρευσε. Και τώρα πάμε στο δεύτερο μέρος της πρωινής συνάντησης, σημαντικό μέρος θα μπούμε ε, στη λίστα των βραβείων Guinness, έτσι, είναι μεγαλύτερος, ο μεγαλύτερος κατάλογος ψηφοφορίας στην ιστορία. Οπότε ελπίζω να είστε έτοιμοι. Ξεκινούμε, ξεκινάμε με ένα τεστ όμως πρώτα μια δοκιμαστική ψηφοφορία, άρχιτη ψηφοφορία. Ψηφίστε παρακαλώ αγαπητοί συνάδελφοι. Πέρας ψηφοφορίας. Πολύ ωραία. Από ό,τι φαίνεται λειτουργεί το σύστημα. Και πάμε στην πρώτη ψηφοφορία, το σημείο 6 της ημερησίας διάταξης. Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που τροποποιεί την ε, οδηγία για την ενεργειακή απόδοση ε, των κτηρίων. Εισηγητής ο κ. Μπέντσεν. Εδώ υπάρχει προσωρινή συμφωνία κατόπιν άτυπου τριλόγου, κανόνας 69F. Έχουμε λοιπόν ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται συγχαρητήρια στο συνάδελφο. Το αποτέλεσμα λοιπόν του τριλόγου θα εξεταστεί στην Ολομέλεια. Πάμε τώρα στην επόμενη ψηφοφορία. Αγαπητοί συνάδελφοι, Παρακαλώ να είστε προσεκτικοί. Θα ψηφίσουμε ε, για το ψήφισμα το οποίο δεν συμφωνεί ε, με την ε, ε πράξη, με τις πράξεις δεξιοδότηση σε ό,τι αφορά την αγορά αερίου. Όποιος είναι κατά του καταλόγου λοιπόν της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πρέπει να ψηφίσει τώρα υπέρ αυτής της αντίρρησης και της μορφής. Όποιος είναι υπέρ όμως της, του καταλόγου της Κομισιόν πρέπει να ψηφίσει κατά της αντίρρησης. Εντάξει. Λοιπόν, άρχεται η ψηφοφορία, ε, ονομαστική προφανώς. Αχά, το ΕΛΚ έχει εδώ δύο μέλη παραπάνω. Όχι, ένα μέλος παραπάνω. Εντάξει, δεν υπάρχει πρόβλημα πλέον. Λοιπόν, απορρίπτεται αυτή η αντίρρηση, αυτή η ε, μομφή. Ο κατάλογος λοιπόν της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, για τα σχέδια κοινού ε, ενδιαφέροντος εγκρίνεται με τις οποίες πράσεις Όλα τα υπόλοιπα ε, πάνε τώρα στον εισηγητή ε, ονομαστική ψηφοφορία επί του κειμένου του συγητή. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ. Πάμε τώρα στο σημείο 9. Α, συγγνώμη. Επί της διαδικασίας. Κάποιος θέλει το λόγο. Παρακαλώ. Σας ακούω. Εκτός μικροφώνου όμως ο μιλητής. Ναι, δεν μπορούσαμε να ψηφίσουμε. Δεν λειτουργήσε το σύστημα. Θα το διορθώσουμε αυτό άμεσα. Ελπίζω να βελτιωθούν τα πράγματα. Στη συνέχεια, ίσως να αλλάξετε θέση. Ή δεν γίνεται αυτό. Εν πάση περιπτώσει θα θα δούμε τι θα γίνει στην επόμενη ψηφοφορία. Εδώ πάντω εμεί ψηφίζουμε υπέρ και στα δύο, οπότε σημειώστε το. Πολύ ωραία, εντάξει. Και τώρα πάμε στην έκθεση της Φρανσουάς ε, Γκροστέτ. Πάλι επί της διαδικασίας θέλει κάποιο λόγο. Ο κύριος Ηλικιώτης, παρακαλώ. Θέλω να σημειώσω από την αρχή όπως προνοεί ο κανονισμός ότι εκ μέρους της GUNGL θα καταθέσουμε άποψη μειοψηφία γραπτός ε, για αυτήν την έκθεση. Ε, και ήθελα να το σημειώσω από την αρχή. Well, uh, do you think on the list of common... Αναφέρεστε στον κατάλογο των σχεδίων κοινού συμφέροντος. Μάλιστα. Την έκθεση για την, ε, που θα μπούμε τώρα σε ψηφορία για το European Defense Industrial Development Program. Η GUNGL θέλει να καταθέσει... Okay θέλει να καταθέσει γραπτό άποψη μειοψηφία. Η οποία βεβαίω είμαστε ενάντια σε αυτήν την έκθεση, αλλά θέλω να καταθέσουμε γραπτό την άποψή μα ω άποψη μειοψηφία. Okay. Notes Okay, Μάλιστα. Πολύ ωραία. Όλα καλά. Αγαπητοί συνάδελφοι, έχουμε πολλές ψηφοφορίες μπροστά μας. Καλό είναι να είμαστε ψύχρεμοι. να μην τρέχουμε όλας να είμαστε ακριβείς και συγκεκριμένοι. Η κυρία Γκροστέτ έχει προετοιμάσει μια έκθεση ε, για τα προγράμματα, για το πρόγραμμα μάλλον ε, ευρωπαϊκής ε, βιομηχανικής ανάπτυξης, αμυντικής ανάπτυξης. Λοιπόν, 35 και 38 μαζί, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 39 του 2007-2008 και άλλα από κοινού 207-208 ενώ ο μελητής υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Συμβασμός 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 2.33 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 2.36 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβασμός 2 και συμβασμός 14α από κοινού υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβασμός 3 και 16 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβασμός 4 και 20 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 269 272 από κοινού 6 τροπολογίες υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 306 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. συμβιβασμός 4α υπέρ κατά να το ελέγξουμε αυτό όμως. 4α. Πολύ ωραία. Ναι, άρχιτη ψηφοφορία. Πάλι έχουμε ένα μέλος του ΕΛΚ που περισσεύει. Ο συντονιστής μας, μάλλον. Ωραία. Πέρας ψηφοφορίας απορρίπτεται. Και πάμε τώρα στο συμβιβασμό 4αα υπέρ κατά να το δούμε και αυτό να το επαληθεύσουμε 4αα έτσι περισσεύει κάποιος από το ΕΛΚ συγγνώμη Πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται λοιπόν. 307 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβασμός 4β υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 308 και 94 από κοινού υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τρεις τροπολογίες από κοινού. 420, 92 και 196 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβασμός 18 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβασμός 5 υπέρ και 21 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Ναι, ναι, θα το επαληθεύσουμε. Γιατί είναι για τον, για τον συμβασμό 5 και 21 λοιπόν, από κοινού. Πέρας ψηφοφορίας, εγκρίνεται. 142 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 14 υπέρ, κατά, αποχές, να το επαληθεύσουμε το, την 14 λοιπόν τροπολογία. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 11 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 341 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 346 και 348 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 44 ε, υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 347 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 350 καθώς και 146 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 18 και 6 υπέρ κατά αποχές α συγγνώμη 18 και 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 349 147 και 45 από κοινού υπέρ κατά να το επαληθεύσουμε αυτό παρακαλώ πέρας ψηφοφορίας απορρίπτεται. 3.52 και 46 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ε, συμβασμός 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 3.90 ε, υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 3.91 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβασμός 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβασμός 8 και 22 υπέρ 23 συγγνώμη 23 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 21 και 187 υπέρ κατά να το επαληθεύσουμε παρακαλώ ψηφίζουμε αυτές τις δύο τροπολογίες από κοινού 421 και 187. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συμβασμός 9. Συμβασμός 10α. Συμβασμός 24. Από κοινού. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβασμός 10 και 25. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνονται. 449 και 189 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 55 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 450 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 448 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Δύο τροπολογίες τώρα. 27 και 12. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δύο τροπολογίες. 451 και 190. Υπέρ. Κατά. Να το επαληθεύσουμε και αυτό παρακαλώ. Δύο τροπολογίες επαναλαμβάνω. 451 και 190. Πέρα τη ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Σαφώ. 191 και 17 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 452 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 453 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 56 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβασμός 11 και συμβιβασμός 26 από κοινού υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 34 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Του συμβασμού 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 52 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβασμός 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 135 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβασμός 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 69 υπέρ κατά να το επαληθεύσουμε. Τροπολογία 69 Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Συμβασμό 15 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβασμός 17 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβασμός 19 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 9 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Και πάμε τώρα στο 114. Στην 114 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 144 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβασμός 22 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβασμός 22α υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 8 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 161 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 163 υπέρ και, 8 από κοινού υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 188 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 206 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 22 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 40 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 42 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 43 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 44 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 37 υπέρ και 1. 37 και 1 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Λοιπόν, τελική ψηφοφορία επί το συνόλου του σχεδίου κειμένου όπως τροποποιήθηκε 52α3 κανόνας, ονομαστική ψηφοφορία, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται σαφώς διαθεσμική διαπραγμάτευση λοιπόν και σχετικός κανόνας 69 γάμα πάλι ονομαστική ψηφοφορία, άρχιτη ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας, έγκριση με μεγάλη πλειοψηφία, συγχαρητήρια στην εισηγήτρια. Και τώρα θα περάσουμε στο επόμενο σημείο. Number 10. Πρόκειται για το σημείο 10. Point number 10 on our um, list of items. Το πέμπτο λοιπόν θέμα, πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την εσωτερική αγορά ηλεκτρισμού. Πρόκειται για recast, στα αναδιατύπωση. Καρίνς είναι ο εισηγητής. Λοιπόν, πρόταση κανονισμού. Πακέτο για την καθαρή ενέργεια. Δεν είναι η πρώτη φορά που ασχολούμαστε με το θέμα αυτό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Ας ξεκινήσουμε. Συμβιβαστική 1. Ποιοι είναι υπέρ κατά αποχές δεκτή. 206 ποιοι είναι υπέρ, κατά, ηλεκτρονικός έλεγχος για την 206. Πέρα της ψηφοφορίας, απερίφθη. Συμβιβαστική 1α ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 1-3-1 και 1-3-2 από κοινού. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος και εδώ παρακαλώ. Κοιτάξτε σε δύο τμήματα. Το πρώτο τμήμα ψηφίζουμε λοιπόν. 1-3-1, τροπολογία 2, πρώτο τμήμα. Πέρα στις ψηφοφορίες. Απερίφθη. Και τώρα περνάμε στην 219. Ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές, ηλεκτρονικός έλεγχος, απερίφθη με την ίδια πλειοψηφία. Περνάμε τώρα στη συμβιβαστική 2. είναι υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. Συμβιβαστική 3. Λοιπόν 286, 287, 288 και 34. Από κοινού. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά ηλεκτρονικός έλεγχος για όλες αυτές. Περνάμε τώρα στην 304. Ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές, απερίφη. Ναι, ήμουν βέβαιος ότι θα ζητήσετε να υπάρξει ηλεκτρονικός έλεγχος. Ψηφίζουμε λοιπόν για την 300... 318... 310, συγγνώμη, υπέρ, κατά, Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 310. Πέρα στις φουφορίες. Απερίφθη. Δεκτή. Προχωράμε. Συμβιβαστική 46. Α, συγγνώμη, 43. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. κάνω λάθη και τα κάνω επίτηδες ηλεκτρονικός έλεγχος. Πέραση ψηφοφορίας. Απερίφθη. 381 και 382. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχέσκα. Πέραση φοφορίας. Δεκτή. Συμβιβαστική 4. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Συμβιβαστική 5. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Ήφησαν. 446 υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 446. Πέρα στις ψηφοφορίες απεριφθήσαν. 447 υπέρ Απερίφθη. Συμβιβαστική 6 ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. Συμβιβαστική 27 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. Συμβιβαστική 4, 24 υπέρ, κατά, για την 45 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 586 υπέρ κατά ηλεκτρονικός έλεγχος 586 ψηφίζεται 224 υπέρ κατά απερίφη Συμβιβαστική 28 υπέρ. Κατά. Αποχές. Αποχές. Απερίφη. Συμβιβαστική 29 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Τέσσερις τροπολογίες τώρα. 2.15, 2.16, 2.17 και 22 μαζί. Ποιοι είναι υπέρ κάτω τροπολογίες λέει ο πρόεδρος, γιατί έχουμε και την έμβη 22 μαζί. Πέρας της ψηφοφορίας. Δεκτή. 2.18 υπέρ κατά. Τι. 5.85, 5.86 και 71 και εδώ ηλεκτρονικός έλεγχος γιατί βλέπω εδώ ότι υπάρχουν διαιρέσεις στο εσωτερικό των πολιτικών ομάδων. 22 β κεφαλαίο περνάμε στη συνέχεια στην 885. 11, 12 και 13. Ηλεκτρονικός έλεγχος. Πέρας της ψηφοφορίας. Συμβιβαστική 25. Ποιοι είναι υπέρ κατά αποχές δεκτή. Κατά αποχές απερίφη. 1119, 1120 από κοινού υπέρ, κατά, αποχές απερίφθησαν. Συμβιβαστική 46 υπέρ, κατά, αποχές δεκτή. 1138 δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Δεκτή. Συμβιβαστική 7 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Συμβιβαστική 8 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Συμβιβαστική 9 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Συμβιβαστική 10 δεκτή. Συμβιβαστική 11 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβιβαστική 12 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβιβαστική 13 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 1256 και NV 119 μαζί πέρας της ψηφοφορίας. Δεκτές. Συμβιβαστική 14. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Ηλεκτρονικός έλεγχος. Πέρα στις ψηφοφορίες. Δεκτή. 15 υπέρ, κατά, αποχές δεκτή. Συμβιβαστική 16 υπέρ, 1348 υπέρ, κατά, αποχές, απερίφθη. 1349 υπέρ, κατά, αποχές, απερίφθη. 1000 μη φορά για την 1351. Πέρα της φοφορίες. Απερίφθη, αποχές, απερίφθη. 1354 υπέρ, κατά, Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 1354. Ψηφίζεται. Πέρας της ψηφοφορίας. απερίφη. Περνάμε τώρα στο 1355. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτό. Δεκτή. Περνάμε τώρα στην 1356 Δέλτα υπέρ. Κατά. Αποχές απερίφθη 1358 υπέρ. Κατά. Αποχές απερίφθη 1359 δι υπέρ. Κατά. Αποχές απερίφθη. Συμβιβαστική 32 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Συμβιβαστική 32α υπέρ. Κατά. 32α ηλεκτρον αποχές δεκτή. Συμβιβαστική 32α υπέρ. Κατά. 32α ηλεκτρονικός έλεγχος. Πέρας της ψηφοφορίας απερίφθη. 33 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Χίλια υπέρ κατά αποχές απερίφθη. Συμβιβαστική 34 υπέρ κατά αποχές απερίφθη. Συμβιβαστική 35 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβιβαστική 36 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβιβαστική 37 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβιβαστική 38 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 1496-1499 υπέρ, κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος για τις δύο τροπολογίες. πέρα της ψηφοφορίας. Απερίφθησαν. 1503 υπέρ, κατά. Αποχές, απερίφθησαν. 1509 υπέρ, πρώτο τμήμα της 1509 υπέρ κατά αποχές απερίφη. συμβιβαστική 39 υπέρ κατά αποχές δεκτή συμβιβαστική 40 υπέρ κατά αποχές δεκτή 1540 υπέρ κατά ηλεκτρονικός έλεγχος για την 1540. ...1541 υπέρ, κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 1541. Απερίφθη για μια ακόμη φορά. Παρακαλώ να σηκώνετε τα χέρια σας. 1542 υπέρ. Κατά. Αποχές απερίφθη 1543 υπέρ. Κατά. Αποχές απερίφθη 1544 υπέρ. Κατά. Αποχές απερίφθη 1545 υπέρ. Κατά. Αποχές απερίφθη 41 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 1546 υπέρ, κατά, αποχές, ηλεκτρονικός έλεγχος για την 1546. Πέρας της ψηφοφορίας. Ένα σοσιαλιστής επιπλέον αυτή τη φορά. Λοιπόν, εντάξει, πέρα τη ψηφοφορία. Απερίφθη. Συμβιβαστική 41α υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 196 υπέρ, κατά, αποχές, απερίφθη. 197 υπέρ, κατά, αποχές, απερίφθη. Τώρα ψηφίζουμε την τροπολογημένη πρόταση, ονομαστική κλίση, ξεκινάει η ψηφοφορία. Ένας επιπλέον από τους σοσιαλιστές, πέρας της ψηφοφορίας. Λοιπόν, ψηφοφορία για να περάσουμε τώρα σε οργανικές διαπραγματεύσεις. Διαδικαστικό. Κάποιος έχει ζητήσει διαδικαστικό πριν την τελευταία ψήφο. Υπάρχει ένα πρόβλημα για την 32α, τη συμβιβαστική αυτή, δεν την ψηφίσαμε, τη για νέο άρθρο, άρα δεν πρέπει να ψηφιστεί. Νομίζω ότι η ίδια άποψη την ίδια απόψη έχει και ο συνάδελφος ε, ο εισηγητής.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 Λοιπόν, αγαπητοί φίλοι, με ηρεμία. Συμφώνησαν ο εισηγητής με τους σκιώδεις ότι θα πρέπει να υπάρξει μία ψηφοφορία όλων των ε, τροπολογιών από κοινού. 116, 137, 139, 705, 177 και 14, 44. Αγαπητοί συνάδελφοι. Είναι πάντα προτιμότερο να διαμαρτύρεστε και να εκφράζεστε όταν υπάρχει ένα θέμα που δεν είναι σαφές. Και αυτό να το κάνετε αμέσως μόλις προκύπτει το θέμα γιατί είχαμε ολοκληρώσει την πρώτη ψηφοφορία και θα ψηφίζαμε το θέμα των διαπραγματεύσεων. Εν πάση περιπτώσει, συμφώνησαν οι εισηγητέ, επανερχόμαστε στην πρώτη ψηφοφορία και ψηφίζουμε τις έξι τροπολογίες από κοινού. Ποιο είναι υπέρ. Κατά αποχές ελέγχουμε ηλεκτρονικά. Ελέγχουμε ηλεκτρονικά. και το αποτέλεσμα είναι τέλος της ψηφοφορίας απορρίπτονται οι έξι τροπολογίες αυτές. Δεν αλλάζει λοιπόν την προηγούμενη ψηφοφορία μας. Το αποτέλεσμα είναι το ίδιο και τώρα αφού ολοκληρώσαμε το τροποποιημένο σχέδιο, C, για τις ε, διαθεσμικές ε, διαπραγματεύσεις. Τέλος της ψηφοφορίας ήταν καθοριστικό αυτό που είπαν. Το θέμα είναι πολύ σημαντικό και για την αγορά της ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και για μας. Η κυρία Νίμπλερ κάτι ότι θα υποβάλω την άποψη της ε, μειοψηφίας για το θέμα αυτό. Oh, he's here. Yes, exactly. Okay. Dear friends, do you need five minute break? break? Χρειάζεται τριών λεπτών. Αλλά τώρα συνεχίζουμε. you uh, You Εχθές ενημερωθήκατε ότι οι τροπολογίες 556, 557 της σελίδας 55, άρθρο 15 και η τροπολογία 622 και 625, σελίδα 56, πρόκειται το άρθρο 16. Αναφέραμε τώρα στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, στην οδηγία για την ηλεκτρική ενέργεια. Θα ψηφιστούν αύριο. Αύριο. Σας ενημέρωσαν εχθές και η ψηφοφορία θα γίνει αύριο. Καταλαβαίνετε, σήμερα είμαστε στο σήμερα και η ψηφοφορία θα γίνει αύριο. Εντάξει, ωραία. Προχωράμε λοιπόν στην επόμενη ψηφοφορία. Πρόκειται για την οδηγία που αφορά τους εσωτερικούς κανόνες για την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Ο εισηγητής είναι ο κύριος Κάρινς. Συμβαστική 19 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 20 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 2.23 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 164 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 2.22 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 2.12 και 2.15 από κοινού υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 208 υπέρ. Κατά. 208 υπέρ. Κατά. Ελέγχουμε την 208. Τέλος. Απορρίπτεται η 208. 209 υπέρ. Με την 224. 209 και 224 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 159 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 132, 28, 217 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 220 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 21 υπέρ. Κατά. Αποχές Εγκρίνεται η συμβαστική 21. 2.38 υπέρ. Το πρώτο τμήμα, το πρώτο. 2.38 πρώτο τμήμα. Κατά αποχές απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 2.47 υπέρ. Κατά. Ελέγχουμε Τέλος. Απορρίπτεται η 247. 33 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Για να ελέγξουμε όμως. Αγαπητοί φίλοι από τους σοσιαλιστές, σηκώστε τα χέρια σας ψηλά. Όχι, ελέγχουμε τη 33 γιατί δεν ήταν σαφές το αποτέλεσμα. Τέλος. εγκρίνεται. 22 συμβαστική υπέρ κατά απόχες υπέρ κατά απόχες εγκρίνεται. Αν δεν ψηφίζετε με σαφήνεια θα κάνω διάλειμμα. Σας παρακαλώ πολύ να είστε προσεκτικοί στο πώς ψηφίζετε. 2,49 υπέρ. Κατά αποχές. Ελέγχουμε τη 2,49. 2,49. Τέλος. Απορρίπτεται. 2,98 υπέρ. Κατά. Ελέγχουμε. Τέλος. Απορρίπτεται. 2,99 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 37 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 38 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 39 υπέρ. Κατά αποχές ελέγχουμε τη 39. Τέλος. Απορρίπτεται 40 υπέρ. Κατά. Ελέγχουμε τη 40. 40. Τέλος. Εγκρίνεται 23 συμβαστική υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 3.10. Κατά. Ελέγχουμε την 310. Τέλος. Εγκρίνεται η 310. Συμβαστική 6. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Οι τρεις επόμενες μαζί. 378. 381 και 49 υπέρ κατά. Τις ελέγχουμε και τις τρεις. Τέλος. Απορρίπτονται. 318, 319 και 42 μαζί υπέρ κατά. Ελέγχουμε αυτές τις τρεις. Τέλος. Απορρίπτονται. 388, 391 υπέρ. Κατά. Ελέγχουμε τις δύο αυτές. Τέλος. Απορρίπτονται. Τέσσερις τροπολογίες μαζί. 3.20 μέχρι την 3.25. Υπέρ. Κατά αποχές, το ίδιο αποτέλεσμα κατά. 3.42, 3.43 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτονται, επίσης απορρίπτονται. 3.44, 3.45 υπέρ. Κατά. Το ίδιο αποτέλεσμα. Κατά. Απορρίπτονται. Τρεις τροπολογίες. 379 μέχρι την 384 υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται. 362, 462 υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται. Συμβιβαστική 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 4, 18 κατά Ελέγχουμε την 418. 418, τέλος, απορρίπτεται. Η 400 και η 401 υπέρ. Κατά αποχές ελέγχουμε, ελέγχουμε. Μάλλον θα απορριφθούν. Τέλος. Απορρίπτονται.

Τέλος. Εγκρίνεται. Συμβαστική 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 4.43 υπέρ κατά αποχές ελέγχουμε. 4.43 έλεγχος. Τέλος απορρίπτεται. 4,59 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ελέγχουμε. 4,59. Τέλος. Εγκρίνεται. 4,54 και 4,56 υπέρ. Κατά. Ελέγχουμε τις δύο αυτές τροπολογίες. Τέλος. Απορρίπτονται. Συμβαστική 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 508. Με 509. Υπέρ. Κατά. Ελέγχουμε. 508-509. Τέλος. Απορρίπτονται. 4.75 το δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Ελέγχουμε. Απορρίπτεται συμβαστική 2 υπέρ κατά αποχές. Εγκρίνεται. 5-23 υπέρ κατά αποχές. Ελέγχουμε. 5-23 λέει ο πρόεδρος. Τέλος. Απορρίπτεται. 3 υπέρ κατά αποχές Εγκρίνεται. 5-5-3 υπέρ. Κατά. Ελέγχουμε την 5-5-3. Ελέγχουμε. Τέλος. Απορρίπτεται. 5-44 υπέρ. Το δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Ελέγχουμε 544. Το δεύτερο τμήμα. Τέλος. Απορρίπτεται με την ίδια πλειοψηφία. 558 έως το 567. Πρόκειται για τέσσερις τροπολογίες υπέρ κατά. Πρέπει να ελέγξουμε 5-5-8-5-6-7. Τέλος. Εγκρίνονται. 5-6-8 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική 4 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δύο τροπολογίες. 6.46 και 6.49 υπέρ κατά απορρίπτονται. 6.18, 6.19, 65 και 6.28 υπέρ κατά αποχές να ελέγξουμε. Τέλος. εγκρίνεται. Τώρα 6.43 υπέρ. Κατά. Πρέπει να ελέγξουμε. 6.43. Τέλος. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 37 για το άρθρο 16α. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Ελέγχουμε. Ελέγχουμε. Δεν είναι σαφές και είναι συμβαστική. Τέλος. Εγκρίνεται. Η συμβιβαστική 33 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται η 33 συμβιβαστική. 7-15 υπέρ και 7-16. 7-15 και 7-16 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτονται. Συμβαστική 9α για την παράγραφο 16. Μάλλον 1-6. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Και τώρα περνάμε σε 8 τροπολογίες. 761 έως την 78 της ένβη που ειναι ταυτόχρονα ταυτόσιμες υπέρ κατά εποχές εγκρίνονται 9β συμβαστική στην παράγραφο 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 7-7-8 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 24 συμβαστική υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 7-9-8 υπέρ. Κατά. Ελέγχουμε. 7-98 ελέγχουμε. Τέλος. Ένας από το ΕΛΚ επιπλέον έχει ψηφίσει. Τέλος της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 7.93 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 25 συμβιβαστική υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 26 συμβαστική υπέρ. Εγκρίνεται 27 υπέρ εγκρίνεται 28 συμβαστική υπέρ κατά εγκρίνεται 29 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 5 5-6 5-5-6 μαζί με την 5-5-7 υπέρ κατά Ελέγχουμε, ελέγχουμε. Τέλος. Απορρίπτονται. Έξι, 22-6-25. Ψηφίζουμε και τις δύο μαζί υπέρ, κατά αποχές. Ελέγχουμε, ελέγχουμε. Μάλλον και αυτές απορρίπτονται. Απορρίπτονται. 30. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 871 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνουμε την 871. Τέλος. Απορρίπτεται. 8.73 υπέρ. Κατά. Ελέγχουμε. 8.73. Τέλος. Απορρίπτεται. 8.74 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Με την ίδια πλειοψηφία. 872, 875 από κοινού υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτονται και αυτές οι δύο. Συμβιβαστική 31 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 32 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 114 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 116 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ναι, ναι, να ελέγξουμε. 116. Τέλος. Εγκρίνεται. με μικρή διαφορά. Συμβαστική 11 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 12 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 13 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 14 συμβαστική υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 6-9 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται ελέγχουμε. Μπορούμε να ελέγξουμε την 969. Το ζητάει ο συντάκτης. Τέλος. Απορρίπτεται. 970. 9.70 υπέρ κατά, αποχές, ελέγχουμε. 971. Κατά, αποχές, απορρίπτεται. 972. Κατά, αποχές, απορρίπτεται. 973. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 15 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 32 συμβαστική. Πέρα. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Η 32 ελέγχουμε. Τέλος της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται η 32. Χίλια υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 1008 υπέρ κατά. Ελέγχουμε την 1008. 1008. Τέλος. Απορρίπτεται. 1007 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 16 συμβαστική υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 1050 έως 1054. 1050 έως 1054, όλες μαζί, πέντε τροπολογίες και ψηφίζουμε υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνονται. 17 συμβαστική υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 1080 υπέρ. Κατά. Εγκρίνουμε. Μα, συγγνώμη, ελέγχουμε την 1080. Τέλος. Απορρίπτεται η 1080. Συμβαστική 18 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 42 και 11, 28 κατά αποχές εγκρίνονται. 43 και 11.30 κατά αποχές εγκρίνονται. 44 και 1131 εγκρίνονται. 1129 κατά αποχές δεν είναι σαφές το αποτέλεσμα. 1129 ψηφίζουμε. Ελέγχουμε ηλεκτρονικά. Τέλος. Εγκρίνεται. Τρεις μαζί. 11.32, 11.33, 11.34. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Ελέγχουμε τις τρεις αυτές τροπολογίες. Τέλος. Απορρίπτονται. Δύο μαζί. 11.35, 11.36. Υπέρ. Κατά. Ελέγχουμε τις δύο αυτές τροπολογίες. Τέλος. Εγκρίνονται. 11.39 υπέρ. Κατά. Ελέγχουμε από κοινού με την 11.40. 11.39 και 11.40. Μα πρέπει να αντιδράσετε. Αλλιώς σημαίνει ότι κοιμάστε, δεν παρακολουθείτε. 11.39 και 11.40 ψηφίζουμε. Τέλος. Απορρίπτονται. 11.41 υπέρ. Κατά. Ελέγχουμε. 11.41. Τέλος. Απορρίπτεται. 34 συμβαστικοί υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. δύο μαζί. 11.52, 11.53. Το δεύτερο τμήμα. Το δεύτερο τμήμα του 11.53 υπέρ. Κατά. Ελέγχουμε. Ελέγχουμε. Τέλος, απορρίπτονται 11, υπέρ. Κατά. Ελέγχουμε. Τέλος της ψηφοφορίας. Απορρίπτω. Κάνουμε τις δύο επόμενες τροπολογίες από κοινού. Ελέγχουμε 1172-1184. Τις δύο από κοινού. Τέλος. Απορρίπτονται. 12.03 υπέρ, κατά. Απορρίπτεται. 12.04 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 12.05. 12.05 έχει αποσυρθεί. Α, έχει αποσυρθεί. Πάμε στη 35 συμβαστική υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 12.42 το πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Απόχες. Εγκρίνεται. 12.42 το δεύτερο τμήμα. Α, θέλετε να ελέγξουμε το πρώτο τμήμα. Εντάξει. Ηλεκτρονικός έλεγχος του πρώτου τμήματος της 12.42. Τέλος της ψηφοφορίας εγκρίνεται. Το δεύτερο τμήμα τώρα, υπέρ, κατά, ελέγχουμε. Μπορεί να έχουμε άλλο αποτέλεσμα. Τέλος. Απορρίπτεται. 12.45 κατά αποχές απορρίπτεται 12.45. 12.45. Έλεγχος. Τέλος. Απορρίπτεται. 12.46 και 12.47. Υπέρ. Κατά. Ελέγχουμε. 12.46-12.47. Ελέγχουμε τις δύο αυτές τροπολογίες. Τέλος. Απορρίπτονται. 12.50 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 12.47 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 12.62 κατά ελέγχουμε την 12.62. Ηλεκτρονικός έλεγχος. Τέλος. Απορρίπτεται. Δύο μαζί. 1268 και 1269. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτονται. Δύο από κοινού. 1272 και 1273. Υπέρ. Κατά. Ελέγχουμε. Πρόκειται για δύο ταυτόσιμες τροπολογίες. Τέλος, απορρίπτεται. Συμβιβαστική 10 από το 1, 2, 3, 4, α και β. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνονται. Λίγες σελίδες α, πιο τα την 131 και την 13 31. Από κοινού. Τέλος της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 13.40 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 13.41 υπέρ. Ναι. Ναι, να ελέγξουμε. 13.40. Εντάξει. Αφού δεν ψηφίζετε, αγαπητοί φίλοι του S&D, ψηφίστε σαφώς. 13.40. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Μικρή διαφορά πάντως. Για μένα έχει απορριφθεί σαφώς βέβαια. Να ψηφίζετε πάντως. 13.41 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 13.42 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 13.43. 13.42. Μάλιστα. 13.42. Επαληθεύουμε. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 13.43. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 13.44. Υπέρ. Κατά. Να το ελέγξουμε. 13.44. Ψηφίζουμε. Πέρας ψηφοφορίας. εγκρίνεται. Τροπολογία 59 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 60 υπέρ. Κατά. Να το ελέγξουμε. Τροπολογία 60 ψηφίζουμε. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 61 υπέρ. Κατά. να το ελέγξουμε. Τροπολογία 61. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 62. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 63. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 64. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 65 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 66 και 3 από κοινού υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 4 υπέρ κατά να το ελέγξουμε. Τροπολογία 4 ψηφίζουμε. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 67 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 68 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 69 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 70 υπέρ. κατά. Να το ελέγξουμε. Ελέγχουμε την τροπολογία 70. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 5 υπέρ. Κατά. Να το ελέγξουμε. Ψηφίζουμε για τροπολογία 5. Πέρας ψηφοφορίας. Α, συγγνώμη εδώ, λάθος δικό μου. Εγκρίνεται. Έχω αρχίσει να πίνω κιόλας. Πάμε πιο κάτω. «117 υπέρ κατά να το ελέγξουμε». Πέρας ψηφοφορίας απορρίπτεται. 72 και 6 από κοινού υπέρ κατά να το ελέγξουμε. Δύο τροπολογίες έτσι. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 71 υπέρ. Κατά. Να ελέγξουμε και την 71. Ψηφίζουμε. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 73 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 75 υπέρ κατά να το ελέγξουμε. Τροπολογία 75. Επαλήθευση. Ψηφίζουμε. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 76 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 77 υπέρ. Κατά. Να το ελέγξουμε. 77. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Συμβασμός 36 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 83 υπέρ. Κατά. Να το ελέγξουμε. Τροπολογία 83. Παρακαλώ. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 85 υπέρ κατά να το ελέγξουμε ξανά. Τροπολογία 85. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται και πάλι. 86 υπέρ. Κατά. Να το ελέγξουμε. 86. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 90 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 91 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 92 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 10 τους ένβη υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 11 υπέρ. Κατά. Αποχές να το ελέγξουμε. Τροπολογία 11. Ψηφίζουμε. Της Envy. Πέρας ψηφοφορίας απορρίπτεται. 98 υπέρ κατά να το ελέγξουμε. 98 ψηφίζουμε. Πέρας ψηφοφορίας απορρίπτεται. 96 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 99 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται και αυτό. 97 υπέρ. Κατά. Να το ελέγξουμε το 97 παρακαλώ. Ψηφίζουμε. Πέρας ψηφοφορίας. Πολύ ωραία. 102 υπέρ. Κατά. Αποχές. Να το ελέγξουμε. 102 λοιπόν. Πέρας ψηφοφορίας απορρίπτεται. 122 υπέρ κατά να το ελέγξουμε και αυτό 122 πέρας ψηφοφορίας απορρίπτεται 121 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 103 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 104 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 105 και 106 από κοινού υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 107 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 110 υπέρ κατά να το ελέγξουμε λοιπόν και αυτό 110 ψηφίζουμε Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 111 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 113 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 112 υπέρ. Κατά να το ελέγξουμε. 112 ψηφίζουμε. πέρα ψηφοφορία απορρίπτεται. 15 υπέρ τη ΕΝΒΗ. Υπέρ. Κατά. Να ελέγξουμε και την τροπολογία 15. Πέρα ψηφοφορία απορρίπτεται. 118 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 119 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 120 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 123 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 124 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 126 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 18 της πέρα. κατά να την ελέγξουμε και την 18 της ΕΝΒΙ ψηφίζουμε πέρας ψηφοφορίας απορρίπτεται και τώρα ψηφίζουμε επί του συνόλου του σχεδίου έκθεσης όπως τροποποιήθηκε ονομαστική ψηφοφορία Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορία. Πολύ ευρία πλειοψηφία. Συγχαρητήρια στον συνάδελφο εισηγητή. Και τώρα ψηφίζουμε για τι θεσμικέ διαπραγματεύσει. Κανόνα 69 69Γ. Ονομαστική ψηφοφορία και πάλι. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Πολύ ωραία. Πάμε λοιπόν για διαπραγμάτευση. Σας ευχαριστώ πολύ. Κύριοι εισηγητές, ε, σκιώδες εισηγητές, ε, θέλω να σας ευχαριστήσω όλους, ε, διότι είχαμε ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. Όλοι οι όλοι οι πραγματικά ήταν εξαιρετικά δραστήριοι. Είχα 18 συναντήσεις με σκιώδεις συγγητές, πρέπει να είναι το ρεκόρ. Αντιλαμβάνομαι ότι δεν είστε έτοιμοι για διάλειμμα. Όχι, όχι, όχι, δεν θέλετε διάλειμμα. Εντάξει, ωραία, δεν κάνουμε διάλειμμα. Και προχωράμε. Αγαπητοί συνάδελφοι, το επόμενο θέμα είναι η ετοιμότητα απέναντι στον κίνδυνο στον τομέα του ηλεκτρισμού, της ηλεκτρικής ενέργειας. Ο κ. Ανωνάτο είναι ο εισηγητής. Τροπολογία 75. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 76. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 77. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 79 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 80 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 81 υπέρ κατά να ελέγξουμε την 81 ψηφίζουμε επί της τροπολογίας 81 81 επαναλαμβάνω Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 82 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 83 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 84 υπέρ. Κατά. Να το ελέγξουμε. 84. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 85 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβασμός 1 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβασμός 2 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 95 υπέρ. Κατά. Να ελέγξουμε. Τροπολογία 95. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Και τώρα ψηφίζουμε ομαδικά 10 τροπολογίες από κοινού. Από την 96 έως την 160 υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται σαφώς. Συμβασμός 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 104 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 105 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται ε, συμβασμός 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται ο συμβασμός 4 109 πρώτο μέρος υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 112 υπέρ. Κατά. Αποχές ε, απορρίπτεται. Συμβασμός 5 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβασμός 6 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 125 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 129 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συμβασμός 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 137 υπέρ κατά αποχές όχι να τσεκάρουμε 137 ελέγχουμε άρχιτη ψηφοφορία πέρας ψηφοφορίας απορρίπτεται δύο τροπολογίες 138 και 139 από κοινού υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 140 υπέρ κατά αποχές γίνεται αποδεκτό. Συμβασμός 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 147 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 148 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 149 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβασμός 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 153 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβασμός 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 15 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 159 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβασμός 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 164 πρώτο μέρος υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 168 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 169 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τρεις τροπολογίες από κοινό 171 173 και 174 υπέρ υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 172 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 175 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 178 υπέρ κατά να ελέγξουμε την 178 την 178 άρχεται ψηφοφορία πέρας ψηφοφορίας απορρίπτεται 179 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβασμός 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 183 υπέρ κατά αποχές α, να το ελέγξουμε 183 ελέγχουμε άρχιτη ψηφοφορία πέρας ψηφοφορίας απορρίπτεται 184 υπέρ κατά να ελέγξουμε και την 184 Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 185 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 186 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 187 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 188 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 189 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 190 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 191 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 192 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 193 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβασμό 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 197 197 υπέρ κατά απορρίπτεται 198 υπέρ κατά εγκρίνεται 198 έτσι ξανά 198 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 199 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 200 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβασμός 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβασμός 15 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 211 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 212 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβασμός 16 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 219 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 220 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 2.21 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 2.22 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 2.23 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 2.24 ε, υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 2.25 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 2.26 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 2.27 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβασμός 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβασμός 17α υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβασμός 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 31 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 35 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 34 α. Όχι, ελέγχουμε την 35. Ψηφίζουμε. 35 πέντε. Πέρας ψηφοφορίας Ναι, ίσως να πρέπει να πάω λίγο πιο αργά. Ε, δεν την κατάλληλη στιγμή. Τότε όμως. Οργανωθείτε καλύτερα. Εγκρίνεται λοιπόν 35 και πάμε τώρα σε συμβασμό 19. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 20. Υπέρ. Συμβασμός 20. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 2. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβασμός 21 υπέρ. 21 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβασμός 24 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβασμός 22 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 52 υπέρ. Κατά να το ελέγξουμε. Τροπολογία 52. Ψηφίζουμε. Πέρας ψηφοφορίας απορρίπτεται. 53 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 54 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβασμός 25 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 58 υπέρ. Κατά. Αποχές να το ελέγξουμε. Τροπολογία 58. Επαλήθευση. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 59 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 59 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 60 υπέρ, κατά, να ελέγξουμε την τροπολογία 60 παρακαλώ. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται 61 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 62 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 63 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 64 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 65 υπέρ κατά να το ελέγξουμε 65 πέρας ψηφοφορίας απορρίπτεται 66 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 67 υπέρ κατά αποχές να ελέγξουμε την τροπολογία 67. Ψηφίζουμε. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται 68 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 69 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 70 υπέρ. Κατά Για άλλη μια φορά παρακαλώ. 70 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται σαφώς. Συμβασμός 23 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 73 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 24 υπέρ. Κατά. Να ελέγξουμε την τροπολογία 24. Α, όχι, είναι σαφώς, απορρίπτεται σαφώς, μάλιστα, απορρίπτεται. 24. Τελική ψηφοφορία. Ονομαστική ψηφοφορία. Φλάβιο Τζανονάτο, ο εισηγητής, πέρας ψηφοφορίας, μεγάλη υποστήριξη, ωραία, και τώρα για τη διαθεσμική διαπραγμάτευση, 69 γάμα 1 Ονομαστική ψηφοφορία. Ψηφίζουμε. Ευχαριστώ. Πέρας ψηφοφορίας. Σαφές το αποτέλεσμα. Συγχαρητήρια, συνάδελφε, Ζανονάτο, καθώς και όλους τους κοιόδους συγκητές. Όλους τους κοιόδους συγκητές. Ευχαριστούμε για τη συνεργασία. Και τώρα ο κύριος Πέτερσεν για το επόμενο θέμα. 86 υπέρ κατά ηλεκτρονικός έλεγχος πέρα στις ψηφοφορίες δεκτή 87 υπέρ κατά ηλεκτρονικός έλεγχος πέρα στις ψηφοφορίες δεκτή. Συμβιβαστική 1 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Μετά περνάμε στην επόμενη σελίδα. 3,99, 96 και 59. Τέσσερις τροπολογίες υπέρ. Κατά. Αποχές απερίφθησαν. 97 υπέρ. Κατά. Αποχές απερίφθησαν. Against. Abstention. Accepted. Compromise 3 in favor. Against. Abstention. Αποχές δεκτή.